Ολοκληρώσαμε το γύρο των ερωτήσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους έλαβαν μέρος στη συζήτηση, υπέβαλαν ερωτήσεις ή παρακολούθησαν την ακρόαση. Ε, πραγματικά ήταν αξιοσημείωτη η τήρηση ε, του, του χρόνου αγόρευσης. Ελάχιστοι βουλευτέ υπερέβησαν το χρόνο ομιλίας τους και σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την πειθαρχία. Ευχαριστώ θερμά και τον ε, υποψήφιο επίτροπο για τις πολύ περιστατωμένες ε, απαντήσεις του και την πληθώρα πληροφοριών που μας έδωσε. Θα ήθελα τώρα να σας υπενθυμίσω μερικά σημαντικά θέματα που ίσως δεν αφορούν άμεσα τη δική μας Επιτροπή Γεωργίας αλλά αφορούν την πολιτική συνοχής στην Ήπεθρο. Πολύ σημαντικό το θέμα της συνοχής ε, στην Ήπεθρο. Κάποια ζητήματα κοινωνικά αφορούν την ε, πολιτική συνοχής και φυσικά επηρεάζουν άμεσα και την Ήπεθρο. Αναφέρθηκε το θέμα του ορίζοντα 2020 και φυσικά η επισητιστική ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια. Άλλοι εξαιρετικά σημαντικοί τομείς. Πολλής λόγος έγινε και για τους εξωτερικούς ε, όρους, την εξωτερική διάσταση και φυσικά την ε, εμπορική πολιτική και την επιρροή της εμπορικής πολιτικής στην γεωργική μας πολιτική. Έχουμε πολύ καλούς ιονούς λοιπόν για τη μελλοντική μας συνεργασία μετά από την πρώτη αυτή ανταλλαγή απόψεων και θα ήθελα να δώσω το λόγο για πέντε λεπτά ακόμη στον υποψηφίο επίτροπο για τα τελικά σχόλια. Αν μπορείτε να κάνετε και μια οικονομία χρόνου, τόσο το καλύτερο. Έχετε το λόγο, κύριε Χόγκαν. Αξιότιμα μέλη. Σας ευχαριστώ για την ευγένεια και την ε, υψηλή ποιότητα των ερωτήσεών σας. Χρειάστηκε να βάλω τα δυνατά μου, αλλά σε ευχαριστώ για τη συνεργασία. Καταλήγοντας, ε, θέλω να καταλάβετε πόσο σοβαρά θα πάρω τα καθήκοντά μου. Η Γεωργία είναι στην καρδιά της ευρωπαϊκής προσπάθειας, είναι μια, ένας τομέας όπου είναι πολύ διαφορετικές οι μέθοδοί μας, τα προϊόντα, η γεωμορφολογία αλλάζουν σε κάθε γωνιά της Ευρώπης αλλά ε, αυτές οι διαφορές είναι η ισχύς της Ευρώπης. Σαν ένα ύφασμα με διαφορετικές πατέντες επάνω του, με διαφορετικά σχέδια επάνω του, είναι μια περιοχή που μας δίνει τεράστιες ευκαιρίες για ανάπτυξη, απασχόληση, για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των αγορών και εντός και εκτός. Πρέπει να αυξήσουμε τις ε, προδιαγραφές μας. Και επειδή οι αναδυόμενες αγορές θέλουν ε, προϊόντα εμπιστοσύνης, η Ευρώπη είναι μοναδική ή μοναδική που μπορεί να τους παράσχει προϊόντα εμπιστοσύνης. Πρέπει λοιπόν να ε, τηρούμε τις προδιαγραφές των οποίων η τήρηση μας κάνει πρωτοπόρους και η αστιφιλία έχει αντιστραφεί εφόσον ε, η παραγωγή τροφίμων γίνεται ιδιαίτερα εξειδικευμένη και υψηλής αξίας δραστηριότητα. Και νομίζουμε ότι έχει επανέλθει και η περηφάνεια των γεωργών, η περηφάνεια στη δουλειά τους, η περηφάνεια ότι είναι σε έναν τομέα που βασίζεται στη φύση και από τον οποίο εξαρτάται η ανθρωπότητα. Και είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Η παραγωγή τροφίμων σε κάθε κράτος μέλος για να ε, ανταποκριθεί στις ανάγκες πρέπει να είναι βιώσιμη. Ο διπλασιασμός της παραγωγής είναι ήδη σημαντικός, αλλά πρέπει να το κάνουμε με τρόπο που να σέβεται την ε, πολυμορφία και τον πλούτο των περιοχών, χωρίς να κάνουμε σπατάλες του νερού που είναι πολύ πολύτιμος πόρος. Και ε, η ενέργεια επίσης πρέπει να καταναλώνεται προσεκτικά και υπό Στην αρχή της θητείας μου θα επισκεφθώ όλα τα κράτη-μέλη Σήμερα είπα πολλά. Όταν όμως θα πάω στα κράτη-μέλη, αντίθετα θα ακούω για να διασφαλίσω ότι η γεωργική πολιτική της Ένωσης θα βασιστεί στον πλούτο της πείρας όλων μας. Η γεωργία πάνω από οποιοδήποτε άλλο τομέα η αντιμετώπιση των ε, σημερινών προκλήσεων θα καθορίσει το μέλλον. Και δεσμεύομαι στα πλαίσια των δυνατοτήτων μου να βασιστώ στην παράδοση, να προωθήσω την κοινοτομία, να εξασφαλίσω ένα μέλλον για την Ευρώπη σε μια νέα παραγωγική και ευημερούσα Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για το κλίμα που επικράτησε στην ακρόαση, για την πολύ καλή διάθεση και τη συμπάθεια που δείξατε. Νομίζω ότι αυτό το φιλικό κλίμα δημιουργεί πολύ καλούς ιονούς για το μέλλον της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαιρόμαστε ιδιαίτερος για την σημερινή μας συνάντηση. Σας ευχαριστώ όλους θερμά, θερμό, θερμά ευχαριστώ και στον Επίτροπο και να σας υπενθυμίσω ότι στις 12.30 σήμερα θα συνεδριάσουν οι συντονιστές και κλεισμένων των θυρών στην αίθουσα ASP 5G3 για την αξιολόγηση. Επαναλαμβάνω 12.30 στην αίθουσα ASP 5 5G3 για την αξιολόγηση. Ραντεβού σε λίγο οι συντονιστές αίθουσα ASP 5G3 στις 12.30. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.